Der Präsident! Meine Damen und Herren, και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ξαναρχίζει η συνεδρίαση. Σας πληροφορώ ότι ο κύριος Ρέστε Ρώση ε, προσθέθηκε στην ομάδα ΕΛΚ από τις 3 Ιουλίου του 2013. Ξεκινούμε με την γεωργία. Ζητήθηκε ονομαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Wir führen diese, we